Well, hello. Hello everyone. Uh, regarding... Καλημέρα σε όλους σας για την ημερήσια διάταξη. Πρέπει να προσθέσουμε ένα σημείο 5 ε, για τον ε, τριμερή διάλογο για τη γενική η νομοθεσία περί τροφίμων. Αν δεν έχετε καμιά επιθυμία για αλλαγή, εγκρίνουμε με, με αυτές τις αλλαγές στην ημερήσια διάταξη και προχωρούμε μέσω στην ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Γκρατσιέλα Γκαβριλέσκου, που είναι αντιπρόεδρο της, της κυβέρνησης της Ρουμανίας και υπουργό Περιβάλλοντος, και τον κύριο Ιωάν που είναι υπουργό υδάτων και Δασών. Θα ήθελα ε, να καλωσορίσω θερμά και τους δύο υπουργού. Καλωσορίσατε στην Επιτροπή μας. Επιευκαιρία, θέλω να συγχαρώ τη Ρουμανία για την πρώτη της Προεδρία του Συμβουλίου και να ευχηθώ στους υπουργού κάθε επιτυχία το ερχόμενο εξάμεινο. Η Ρουμανική Προεδρία θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο γιατί θα κληθεί να κλείσει μια σειρά σημαντικών θεμάτων ε, που ε, εμπίπτουν στη δική μας αρμοδιότητα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σε λίγες εβδομάδες ουσιαστικά από σήμερα ε, και έχουν προγραμματίσει και πολλές εκδηλώσεις υψηλού ενδιαφέροντος για μας, μεταξύ αυτών κλιματική αλλαγή, διαχείριση των υδάτων, βιοπικιλότητα και βιώσιμη ανάπτυξη. Όσοι ήθιστε, στην αρχή της Προεδρίας, η Αντιπρόεδρος και ο Υπουργός θα μας παρουσιάσουν τις βασικές προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας για το περιβάλλον και το κλίμα και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής μας. Τούτων όλων λεχθέντων περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ έχετε το λόγο. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, Αγαπητά μέλη, καταρχήν σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να συμμετάσχω σε αυτή την παραδοσιακή συνάντηση που λαμβάνει η χώρα στην αρχή κάθε προεδρίας, εκπεριτροπής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και θα ήθελα να συνεχίσουμε αυτό το διάλογο μαζί σας και κατά το επόμενο εξάμεινο. Πιστεύω πιστεύω ότι ο διάλογος και η συνεργασία μας θα πλαισιώσει τις προσπάθειες που θα πρέπει να αναλάβουμε και ξεχωριστά αλλά και μαζί για να δώσουμε τελική μορφή στις διαπραγματεύσεις για το νομοθετικό μας έργο. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα που είναι περιορισμένο, είμαστε πεπισμένοι ότι από κοινού θα μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε τις σημαντικότερες και καλύτερες λύσεις για την ευρωπαϊκή ατζέντα. Η Ρουμανία αναλαμβάνει για πρώτη φορά την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και θα ήθελα να σας τονίσω ότι θα αναλάβουμε κάθε προσπάθεια ε, και θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το έργο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Βασιζόμαστε βεβαίως στα κράτη-μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε στη συνέχεια να σας παρουσιάσω εντάχει τις προτεραιότητες και τους στόχους της ε, Ρουμανικής Προεδρίας στον τομέα των κλιματικών αλλαγών και της προστασίας του περιβάντος. Έχουμε να δράσουμε μέσα στα, σε τέσσερις ε, πυλώνες. Σε την Ευρώπη της σύγκλησης, την Ευρώπη της ασφάλειας, της Ευρώπης ως ε, παγκόσμιο δράστη και της Ευρώπης για τις κοινέ αξίες. Οι κλιματικές αλλαγές εντάσσονται στα πλαίσια του πυλώνα της Ευρώπης της σύγκλησης, λαμβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Ατζέντα αλλά και τη Διεθνή Ατζέντα, η Ρουμανική Προεδρία θα λάβει υπόψη τις κλιματικές αλλαγές, την βιοπικιλότητα, την βιώσιμη ανάπτυξη και την διαχείριση των υδάτων. Το τελευταίο θέμα περί διαχείρισης των υδάτων θα παρουσιαστεί από τον Υπουργό Δασών και Υδάτων Ντένες. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στα εξής. Η Προεδρία θέλει να δώσει τελική μορφή στο θέμα που αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος για τα βαρέα οχήματα. Αυτό, αυτή είναι και η ψηφίδα που λείπει σε σχέση με τα μέτρα μείωσης εκπομπών διοξιδίου άνθρακα στον τομέα των οδικών μεταφορών. Η εφαρμογή αυτού του κανονισμού θα αποτελέσει σημαντική συνεισφορά στην των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ε, κλιματικές αλλαγές και για την μείωση των εκπομπών σε εθνικό επίπεδο με βάση του κανονισμού περί επιμερισμού προσπαθειών. Πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε εν ευθέτω χρόνο σε μία συμφωνία σε σχέση με τον κανονισμό αυτό, ο οποίο θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή πριν από το τέλος τη θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ρουμανική Προεδρία θα προωθήσει και το νέο πρόγραμμα LIFE για την χρηματοδότηση του περιβάλλοντος και των δράσεων στον τομέα του κλίματος. Θεωρούμε ότι θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση καθώς και άλλες οριζόντιες πτυχές μετά από τη Συμφωνία Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ρουμανική Προεδρία αναμένει με ενδιαφέρον τις διαπραγματεύσεις διαπραγματεύσεις, τις επικοδομητικές διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το σημαντικό θέμα. Παράλληλα, αναμένουμε και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κανονισμό που αφορά τον μηχανισμό επαλήθευσης και δράσης όσον αφορά την, ε, τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Η Ρουμανική Προεδρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να προωθηθούν αυτά τα θέματα το ταχύτερο δυνατόν. Επίσης, θα ασχοληθούμε και με τις δημόσιες συζητήσεις σε επίπεδο Συμβουλίου για ένα κοινό όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μακροχρόνια στρατηγική όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές καθώς και μια βιώσιμη, ένα βιώσιμο μετασχηματισμό της οικονομίας. Οι συζητήσεις θα είναι ολοκληρώσεις έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ιδιαίτερα οι Ευρωπαίοι πολίτες, να προωθήσουν αυτό το πρότυπο ανάπτυξης. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Μιλάμε για την απομάκρυνση από τον άνθρακα και τη βιωσιμότητα που αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη αλλά και για τον πλανήτη καθώς και για την οικονομική ανάπτυξη και τον εργασιακό χώρο κατά τις επερχόμενες δεκαετίες. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η διαδικασία ε, μετασχηματισμού δεν θα αφήσει απ' έξω καμία περιφέρεια και κανέναν πολίτη. Η, η προστασία της βιοπικιλότητας είναι μία από τις προτεραιότητες μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 23% της επιφάνειας των χωρών αφορά υδάτινους πόρους, καθώς και φυσικούς πόρους που την χάνουν προστασία από το Natura 2000. Μέσα στα πλαίσια της COP14 θα λάβουμε υπόψη και την ε, ε, βιολογική ποικιλότητα και θα ολοκληρώσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις ενώ της COP15 το 2020 στο Πεκίνο και μέσα στα πλαίσια της βιοπικιλότητας 2011-2020 και για την βιοπικιλότητα βιοπικιλότητα μετά το 2020. Υπ' αυτή την έννοια θα οργανώσουμε στο Βουκουρέστι το Μάιο στα πλαίσια του άτυπου Συμβουλίου Περιβάλλοντος μία συζήτηση επί του θέματος και ελπίζουμε τα αποτελέσματα αυτών των συζητήσεων να αποτελέσουν σημαντικά να δώσουν σημαντικά μηνύματα και να αντλήσουμε διδάγματα σε σχέση με την βιοποικιλότητα μετά από το 2020. Επίσης, μας απασχολεί το θέμα του ψηφίσματος αφορά, που αφορά την COP14. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις οικολογικές σχέσεις που ορίζουν το φυσικό περιβάλλον. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μια σωστή προσέγγιση ως προς τη διαχείριση των φυσικών πόρων και γι' αυτό στο Φουκουρέστι στις 6 και 7 Ιουνίου θα ασχοληθούμε με, θέμα, με το θέμα της διαχείρισης των ε, μεγάλων σαρκοβόρων προκλήσεις και λύσεις. Επίσης, θα μας απασχολήσει και το θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ιδιαίτερα ο δεύτερος κύκλος για την αναθεώρηση των νομοθετικών μέσων για το περιβάλλον. Θα οργανωθεί μία πολιτική ε, συζήτηση, μια συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο για τους για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν θα προβάλλουμε συγκεκριμένα φιλόδοξα μέτρα για να μειώσουμε την έκθεση και στους χημικούς παράγοντες. Προσδίδουμε μεγάλη σημασία στο περιβάλλον και στην βιώσιμη ανάπτυξη θεωρούμε ότι το περιβάλλον ε, είναι ε, η κινητήριος δύναμη της πράσινης ανάπτυξης και ενθαρρύνει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Γι' αυτό και θα πρέπει να παγιοποιώσουμε αυτό το τομέα. Η Ρουμανική Προεδρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια μέσα στα πλαίσια της τέταρτης συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ούνεα 4, που θα λάβει το Μάρτιο στο Ναϊρόπι. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις ε, προκλήσεις υπέρ του περιβάλλοντος καθώς και τα βιώσιμα μέτρα και σχήματα κατανάλωσης. Παράλληλα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που προσδίδουμε στην εφαρμογή της Ατζέντα 2030 για την βιώσιμη ανάπτυξη στις 16 Απριλίου του 19 θα οργανωθεί στο Βουκουρέστι η Διεθνής Διάσταση διάσκεψη Ατζέντα 2030 εταιρικέ σχέσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη. Λαμβάνοντας υπόψη και το Παγκόσμιο Σύμφωνο Περιβάλλοντος, θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε και νομικά, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα διεθνή μέσα υπέρ του περιβάλλοντος που μας ενισχύουν. Παράλληλα με την ΟΥΝΕΑ, η Ρουμανική Προεδρία θα συμμετάσχει σε όλες τις ε, θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης τις διεθνείς συναντήσεις που προβλέπονται. Η 8 διάσκεψη συμβαλωμένων μερών στο ΕΣΠΟ ΜΟΠ 8 στη Γενέβη 5 7 Φεβρουαρίου. Τριμερής διάσκεψη στον τομέα της αντιμετώπισης των αποβλήτων και των χημικών ουσιών στην Βασιλεία, Ρότερνταμ και στο Χόλμη στις 29 Απριλίου μέχρι 10 Μαΐου. Επίσης, την 7η σύνοδο των ε, διακυβερνητικών πλατφορμών για την βιοπικιλότητα στο Παρίσι 29 Απριλίου με 4 Μαΐου, καθώς και την διάσκεψη ΣΥΤΕΣ στη Σρι Λάνκα από τις 23 Μαΐου μέχρι τις 3 Ιουνίου και την διάσκεψη διεθνών ε, διαπραγματεύσεων για τις κλιματικές αλλαγές στη Βόνη από τις 17 μέχρι τις 27 Ιουνίου. Τέλος, θα ήθελα να σας τονίσω ότι είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε από κοινού για να αντιμετωπίσουμε τις κοινέ προκλήσεις, γιατί για πρώτη φορά αναλαμβάνουμε αυτό το ρόλο, αλλά θεωρώ με μεγάλη ευθύνη και οριμότητα. Πρόκειται για ε, ένα μέσο το οποίο μετερχόμαστε μέσα στα πλαίσια το οποίο μετερχόμαστε μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας. Για να φτάσουμε σε αίσιο πέρας θέλουμε άμεσο διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς έτσι ώστε να δούμε κάθε πτυχή κοινού ενδιαφέροντος σε σχέση με την ευρωπαϊκή ατζέντα για να δούμε ποιες είναι οι ενδεχόμενες λύσεις. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στο γεγονός ότι οι προσπάθειες μας θα αποτελέσουν προστιθέμενη αξία στις προγενέστερες προεδρίες σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Επιτροπή για να φτάσουμε σε λύσεις σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις. Εμείς μιλάμε για την συνοχή, την κοινή αυτή ευρωπαϊκή αξία που αποτελεί προτροπή έτσι ώστε να δώσουμε μεγάλη η μάχη υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Το λόγο έχει ο Υπουργός Δένες, ε, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις προτεραιότητες στον τομέα των ε, υδάτων και των δασών. Αξιότιμη Πρόεδρε, κύριοι Ευρωβουλευτές, η Ρουμανία στα πλαίσια της Προεδρίας θα υποστηρίξει τις ε, προσπάθειες έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ακόμα πιο δυνατή και ακόμα πιο δυναμική. Η διαχείριση των υδάτων είναι ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος και η πρόθεση των διαπραγματεύσεων για αυτά τα δύο θέματα αποτελεί άμεση προτεραιότητα στα πλαίσια της Προεδρίας μας. Σας το αναφέρω αυτό γιατί η οδηγία που αφορά το πόσιμο είδωρ αφορά την ποιότητα των υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρχική οδηγία εγκρίθηκε εδώ και 20 χρόνια και αυτή η πρόταση προβλέπει την βελτίωση συγκεκριμένων πτυχών σε σχέση με το REFIT, καθώς και την ενημέρωση των παραμέτρων, των ποιοτικών παραμέτρων, με βάση την αναγνώριση κινδύνων, το διαχειριστικό πλαίσιο, την εναρμόνιση των προτύπων καθώς και την βελτίωση της ποιότητας του ύδατος. Η Βουλγαρική καθώς και η Αυστριακή Προεδρία κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες έτσι ώστε να γίνουν καλές διαπραγματεύσεις. Η Ρουμανική Προεδρία θα προωθήσει αυτό το θέμα ακόμα περαιτέρω. Ήδη από τις αρχές του Ιανουαρίου έχουμε τρεις συναντήσεις των ομάδων εργασίας και πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε σε βελτίωση όλων των τεχνικών πτυχών. Θα συνεχίσουμε με αυτό τον επιταχυμένο ρυθμό εργασιών. Θα Ευχαριστούμε μαζί σας ε, την αμέσως επόμενη περίοδο για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ανοίξουμε τις διαπραγματεύσεις. Η βασική μας προτεραιότητα είναι να φτάσουμε σε ένα εξισορροπημένο συμβαστικό κείμενο για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος που να μην επαυξάνει το κόστος που να επιβαρύνει τους πολίτες. Επίσης, το υδάτινο έλλειμμα πλήττει το 1 τρίτον της εδαφικής επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν αφορά μόνο τον Νότο. Η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων αποτελεί μια εναλλακτική πρακτική λύση έτσι ώστε να ε, έχουμε ένα αποδοτικό πλαίσιο μέσα στα πλαίσια της ε, κυκλικής οικονομίας. Το Μάιο του 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μία πρόταση κανονισμού για τις ελάχιστες προδιαγραφές χρήσης υδάτων για την άρδευση. Μιλάμε για μια κοινή προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις για να υπάρχει συνάφεια και προβλεψιμότητα για τους επενδυτές που θέλουν να επαναχρησιμοποιήσουν τα ύδατα. Η Ρουμανική Προεδρία θα προωθήσει αυτό το θέμα με μια πολιτική συζήτηση στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος. Και αυτό θα γίνει ήδη από τον Μάρτιο λοιπόν να έχουμε μία καλή προσέγγιση για το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος στον Ιούνιο. Αναμένουμε τις εξελίξεις και τη δική σας συνεργασία. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική αποτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με με το κανονιστικό πλαίσιο στον τομέα των υδάτων, καθώς και οι συζητήσεις σε διεθνές επίπεδο για τους στόχους της Ατζέντα 2030 σε σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον, μετά από την άτυπη συνάντηση του Συμβουλίου, στις 21 και 22 Μαΐου του θα γίνει μία διεθνής διάσκεψη στο Βουκουρέστι. Ε, αναμένω τις ερωτήσεις σας και ελπίζω να μπορέσω να ανταποκριθώ με τις απαντήσεις μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφοι, ο συνήθως, καλό καταρχήν και τους συντονιστές ή τους αντικαταστάτες τους να πάρουν το λόγο δύο λεπτά ο καθένας ή η καθεμία και μετά θα απαντήσουν οι δύο προσκαλισμένοι υπουργοί για να ακολουθήσει ένα δεύτερος γύρος ομιλητών με ένα λεπτό ε, για τον καθένα. Ο κ. Λίζε καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους δύο υπουργού, την κυρία Προεδρεύουσα και τον κύριο Προεδρεύοντα. Δύο σημεία θέλω να αναφέρω. Το είναι η προστασία του κλίματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είπατε και εσείς, κατέθεσε τις ιδέες της για μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική μέχρι το 2050. Προσωπικά και νομίζω ότι μπορώ να μιλήσω και εξ ονόματος πολλών παρόντων συναδέλφων. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική αυτή την παρουσίαση ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας σε συνεργασία με τον Πρόεδρο Τούσκ του Συμβουλίου να επιληφθεί του κειμένου αυτό το Συμβούλιο και δυνατόν και στη Σύνοδο Κορυφής για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Συμπίου να αποφασίσει μια ε, στρατηγική για το τι θέλει να κάνει με την προστασία του κλίματος και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αυτά χρειάζονται και μια προετοιμασία σε υπηρεσιακό επίπεδο. Πώς ε, το βλέπετε πριν τα συζητήσει το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το δεύτερο αφορά την καθαρή ατμόσφαιρα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει προόδους ε, για τα σωματίδια της χώνης και τα ε, οξύδια του αζότου. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο στόχο που είχαμε θέσει βέβαια, αλλά γίνεται μια πολύ έτσι, επικριτική συζήτηση αν είναι σωστέ οι αριακές τιμέ που έχουμε θέσει. Εσείς την παρακολουθείτε ε, αυτή τη συζήτηση, την επιστημονική, την έχετε παρακολουθήσει και πώς έχετε αντιδράσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η ε, κυρία Ντάλη. Eh, Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τις δύο, τους δύο υπουργού. Χαίρομαι που είστε εδώ ενώπιόν μας και μας παρουσιάζετε τις προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας στα θέματα περιβάλλοντος. Καλωσορίζουμε αυτές τις προτεραιότητες, τις χαιρετίζουμε. Ιδιαίτερα η δική μου κοινοβουλευτική ομάδα υπό την ε, προεδρία σας βρισκόμαστε στο τελευταίο κομμάτι της θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώπιον ενό Brexit κλπ. κλπ. Η συγκυρία είναι περίπλοκη. Θέλω να εστιάσω σε μια-δύο από τι προτεραιότητε αυτές για να σα ζητήσω περισσότερε πληροφορίε για το πώ σκοπεύετε να πετύχετε του στόχου σας, τους στόχους αυτούς που έχετε εσείς ίδιοι θέση. για την ε, νέα διευκόλυνση συνεδέοντας την Ευρώπη. Είπατε ότι θα δημιουργηθεί ε, ένα ταμείο για τα εναλλακτικά κάψιμα, ιδιαίτερα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θα μπορούσατε να μου δώσετε λίγο περισσότερες πληροφορίες για αυτό το ζήτημα. Για αυτές τις δύο προτεραιότητες. Επίσης είπατε ότι θα γίνει μια συζήτηση για την είναι η θέση περιπτή ε, στα στρατηγικών σχεδίων για τις μπαταρίες. Είπατε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι ηγέτη σε ό,τι αφορά ε, τους συσσωρευτές και την αποθήκευση ενέργειας. Πώς σκοπεύετε να προχωρήσετε με αυτό το θέμα. Η... Επίσης, η Προεδρία, είπατε, θα εστιάσει στην ε, μείωση της, ε, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα νέα βαρεοχήματα. Δεν ξέρω πόσο επίμαχα είναι αυτά τα θέματα στο Συμβούλιο. Τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές και διστάμενες απόψεις. Ελπίζω όμως ότι η Ρουμανική Προεδρία θα καταφέρει να προχωρήσει. Πριν κλείσω, θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που το Συμβούλιο υιοθέτησε το συμβιβασμό για τα ελαφρά οχήματα. Η Προεδρία κατάφερε εξασφαλή συμφωνία. Συγχαρητήρια. Πρόεδρος, ο κ. Ντεμέρσμακερ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί Υπουργοί, καλωσορίσατε ορίσατε θερμά εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ως πρώην εισηγητής για τη βιοποικιλότητα και την αντίστοιχη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεωρώ πολύ σημαντικά τα θέματα της φύσης και της βιοπικιλότητας. Είναι πολύ ψηλά και στις δικές μου προτεραιότητες και είμαι βέβαιος και στις δικές σας. Και η ίδια η Ρουμανία είναι θησαυρό από βιοπικιλότητα. Ε, στα Καρπάθια βλέπουμε ε, μια πραγματικά παρθένα φύση από τις τελευταίες εκατοντάδες μοναδικά φυτά για την Ευρώπη και πολλά σαρκοφάγα, λύκους, αρκούδες και λίγκες ακόμα. Αλλά στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και στον υπόλοιπο κόσμο δυστυχώς δεν είναι τόσο ωραία αυτή η εικόνα. Κυρία Υπουργέ, ο προκάτοχός σας στη ρουμανική κυβέρνηση ε, τώρα είναι διευθυντής, διευθύντρια μάλλον ε, στην αντίστοιχη επιτροπή του ΟΗΕ για τη βιοπικιλότητα και είπε ε, πρόσφατα στην Αίγυπτο ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με τη βιοπικιλότητα και ε, την καταστροφή των ειδών γιατί σε λίγο θα χτυπήσει η καμπάνα για την καταστροφή του ίδιου του ανθρώπου. Ε, πραγματικά είναι μια κρίση κλιματική αυτή που γνωρίζουμε και πηγαίνουμε προς την καταστροφή. Ε, ε, υπάρχουν διάφορες εκθέσεις, ένας δείκτης Living Planet. Ποτέ δεν έχουμε χάσει τόσα πολλά άγρια ζώα. 60% είναι λιγότερη σήμερα η άγρια πανίδα σε σχέση με 40 χρόνια πριν και ε, ε, είναι ανθρωπογενείς οι παράγοντες μεταξύ άλλων υπεραλίευση, αλλαγή του κλίματος κτλ. Είναι πραγματικά η ανθρώπινη δραστηριότητα που προκαλεί αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει ε, να παραμείνει σε μια έξυπνη και βιώσιμη Ευρώπη προτεραιότητα η επένδυση στη βιοπικιλότητα. Και σας ερωτώ, βεβαίως έχει σημασία να υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη στη μετάβαση προς μια οικονομία μια βιώσιμη και ε, κυκλική και με λιγότερο δεξίδι του άνθρακα. Αυτό κάνει και το πρόγραμμα LIFE, το είπατε κι εσείς. Ε, τα έργα του LIFE είναι ένας μοχλός που μπορεί να βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό προς την κατεύθυνση αυτή. Οι επενδύσεις από το LIFE είναι ε, κρίσιμες και για τη φύση και για τον άνθρωπο. Ακούω λοιπόν ότι θέλετε να κάνετε και μεγάλες πρόοδους στις διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα LIFE. Μήπως μπορείτε να μας τα πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα, με περισσότερες ε, λεπτομέρειες, τι σημαίνει σημαντική πρόοδος. Υποστηρίζετε το κοινοβούλιο ε, που ζητάει περισσότερα χρήματα για το live. Και επίση, ποια είναι η θέση σας απέναντι στο αίτημα για περισσότερη συνάφεια και συνοχή μεταξύ των διαφόρων ε, ταμείων βλέπε live Ταμείο Συνοχής και Ταμείο για τη Γεωργία. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Now, Mr. Gerbrandi. Ευχαριστώ κύριος στα αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ τους δύο υπουργούς που βρίσκονται στο δικό μας εδώ τροπικό οικοσύστημα, στο Κοινοβούλιο. Με χαρά τους ε, υποδεχόμαστε. Δύο θέματα θέλω να θίξω. Πρώτον, η μακροπρόθεσμη κλιματική στρατηγική για το 2050. Κρίσιμο σημείο, όχι μόνο για το ίδιο το κλίμα, αλλά και για την οικονομία. Αν δείτε τα νούμερα, τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία προέρχονται από τις ε, ε, ε μελέτες της Κομισιόν, αναφέρουν ότι θα μπορούσαμε να από να εξοικονομήσουμε μέχρι το 2050 2-3 εκατομμύρια ευρώ από την ε, ε, για, από τους ενεργειακούς πόρους. Τεράστιο ποσό. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Κεντρικές ε, Τράπεζες επίσης προειδοποιούν για κινδύνους που, που συνδέονται με το κλίμα και υπογραμμίζουν τη σημασία να έχουμε σαφάνεια, σαφήνεια και διαφάνεια μακροπρόθεσμα για τις επιχειρήσεις ό,τι αφορά το περιβάλλον και την ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι δεν θέλουμε απλώς ε, ε, ε μια ισχυρή θέση από το Συμβούλιο για τη στρατηγική μέχρι το 2050, αλλά θα πρέπει να αλλάξουμε και τους στόχους για το 2030. Οπότε η ερώτηση μου είναι τι θα γίνει στο Συμπίου, στην ε, εκτακτή διάσκεψη κορυφής, ε, στο εκτακτό ε, ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε σχέση με αυτό το θέμα. Μετά, βιοπικιλότητα. Δεν θα επαναλάβω τα όσα είπε ο κ. Ντεμέρσμακερ, αλλά θέλω να υπογραμμίσω τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου του 2018, όπου το Συμβούλιο αναφέρει, καλεί την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να αυξήσουν τις δράσεις τους τα επόμενα δύο χρόνια για να αντιμετωπίσουν τις βασικές αιτίες της μείωσης της, ε, της απώλειας βιοποικιλότητας και να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ε, τα εθνικά σχέδια υπέρ της βιοποικιλότητας και την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα μέχρι το 2020. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να ε, εντείνουμε τις προσπάθειές μας υπέρ της βιοποικιλότητας. Χρειαζόμαστε, χρειάζεται να κάνουμε πολύ περισσότερα από ό,τι στο παρελθόν. Δεν είναι δυνατόν η, η, η, η στήριξη της βιοπικιλότητας να γίνεται ε, μεμονωμένα, κατακαιρματισμένα, χωρίς να συνδέεται και με άλλες πολιτικές, όπως για παράδειγμα την κοινή αγρογεωργική πολιτική. Θα μπορούσατε εσείς να μας πείτε ποιοι είναι οι στόχοι σας για τους επόμενους μήνες, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για το 2020. Ο κ. Σέικχαουτ. Uh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τους υπουργούς για την εισαγωγή τους. Ήταν ε, χαρά μου την προηγούμενη εβδομάδα να συμμετάσχω στον πρώτο τριμερή διάλογο ε, της ε, Ρουμανίας για τα βαρέα οχήματα και το διοξείδιο του άνθρακα βάπτισμα πυρός για την Ρουμανική Προεδρία. Ε, ελπίζω ότι ε, θα προχωρήσουμε εκεί. Το Συμβούλιο θα πρέπει να μετακινηθεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά εν πάση περιπτώσει εμπιστεύομαι την Ρουμανική Προεδρία. Να σχολιάσω κάποια πράγματα που είπαν και οι προηγούμενοι. Για παράδειγμα, για το κλίμα, για την μακροπρόθεσμη στρατηγική δεν έχουμε μόνο τη σύνοδο κορυφή του Συμπίου, ε, αλλά και το τι θα, ποια θα είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ περιμένει προσδοκά από τους και κρατών κυβερνήσεων να κάνουν περισσότερα πράγματα και ότι και η Ευρώπη έχει μείνει πίσω. Ιστερεί. Οπότε, τι πρόκειται να κάνει η Ρουμανική Προεδρία έτσι ώστε η Ευρώπη να μην πάει με άδεια χέρια το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν οδυνηρό τουλάχιστον. Δεύτερον, για τον Υπουργό. Ε, Μιλήσατε για την οδηγία μου Δεν Δίδατος είναι σημαντικό θέμα, το καταλαβαίνω γιατί δίνετε πρωτοβουλία, κύριε Τένες. Ε, τι θα κάνετε όμως έτσι ώστε η θέση του Συμβουλίου να συγκλίνει με τη θέση του Κοινοβουλίου ε, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πολύ μακριά από τη δική μας θέση. Ποια είναι η δική σας σε αυτό το θέμα. Και δύο ακόμα θέματα που έχουν σχέση με την συνέπεια και συνέχεια ε, θεμάτων τα οποία έχουν περιβαλλοντικές διαστάσεις δεν είναι όμως απόλυτα ε, περιβαλλοντικά. Για παράδειγμα, η βιώσιμη χρη, χρηματοδότηση δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά και περιβαλλοντικό θέμα. Το θέμα δεν είναι να ορίσουμε τι είναι βιώσιμο αλλά να ορίσουμε και τι είναι μη βιώσιμο στην οικονομία. Και μετά η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Ξέρω ότι ο Υπουργό ε, Γεωργίας Γεωργίας θα είναι εδώ αύριο, θα το συζητήσουμε μαζί του, αλλά είναι πολύ πολύ σημαντικό να το δουν και οι Υπουργοί Περιβάλλοντος. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι το Συμβούλιο Περιβάλλοντος θα συμμετάσχει πλήρως στην συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Εδώ κλείνουμε λοιπόν η πρόεδρος τον πρώτο γύρο ομιλητών. Σας καλώ τώρα να απαντήσετε στον πρώτο γύρο των ερωτήσεων. Η κυρία Γκαβριλέσκου έχει πρώτα το λόγο και στη συνέχεια ο κύριος ε, Ντένες θα μπορούσε να συμπληρώσει ενδεχομένως Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, ερωτήσεις σας και σας λέω εξ αρχής ότι όλα τα θέματα που θίξατε είναι ύψης της σημασίας και για η Ρουμανική Προεδρία και όπως σας υποσχέθηκα εξ αρχής, θα ασχοληθούμε με όλες τις προτεραιότητες εκ του σύνεγγης, έτσι ώστε να προωθηθούν όλες οι διαπραγματεύσεις και να να τις ολοκληρώσουμε. Ο κύριος ε, Λίζε μίλησε για μία ανησυχία που είναι κοινή μας ανησυχία. Πρόκειται για την μακροχρόνια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κλιματικές αλλαγές. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και οφείλω να σας πω ότι η Ρουμανική Προεδρία θα προωθήσει συζητήσεις σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο, όπως και πρέπει, όχι μόνο μέσα στα πλαίσια του Συμβουλίου Περιβάλλοντος αλλά και γεωργίας, ανταγωνιστικότητας, ενέργειας και μεταφορών. Σε όλα αυτά τα συμβούλια. Και θα αναλύσουμε τις δυνατότητες που δια γράφονται με βάση αυτή τη συζήτηση και σε επίπεδο ΕΚΟΦΗΝ ως προς το εργατικό δυναμικό. Μιλήσατε για την διάσκεψη στο Σιμπίου το Μάιο όπου εμείς αλλά και ολόκληρος ο κόσμος θα συνεισφέρει και θα αποτελέσει ένα θετικό βήμα για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής ως προς τις ε, κλιματικές αλλαγές μακροχρόνια. Κύριε Λίζε, όλοι συμφωνούμε ότι πρόκειται για τον κύκλο ζωής του πλανήτη μας. ως προς την ε, ποιότητα του αέρα και των υδάτων. Αυτά είναι ζητήματα που άπτονται του του περιβάλλοντος, της πολιτικής περιβάλλοντος και εμείς ως Προεδρία αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνδράμουμε όπως ακριβώς και η Επιτροπή. Θα πρέπει να κάνουμε μία προβολή προς το μέλλον. Αυτό κάνει και η Επιτροπή. Έχουμε μία αξιολόγηση της Επιτροπής σε σχέση με τις οριακές ε, τιμές της Κομισιόν και από την ποιότητα του αέρα εξαρτάται και η ζωή των πολιτών, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά ανά τον κόσμο. Κυρία Ντάλη, ήταν πολύ διορατική η ερώτησή σας όταν μιλάμε για καθαρά οχήματα και για απομάκρυνση από τον άνθρακα, θα πρέπει να προτείνουμε προγράμματα και σχέδια που να μπορέσουν να εφαρμοστούν σε ευρεία κλίμακα, ξεκινώντας όμως από μία περιορισμένη κλίμακα, δηλαδή των τοπικών αρχών, μέχρι το πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σε σχέση τώρα με την αναθεώρηση της οδηγίας για τα καθαρά οχήματα, αυτή η οδηγία είναι προτεραιότητά μας. Μιλάμε για καθαρά οχήματα και όταν λέμε καθαρά μιλάμε για μείωση των ε, ρήπων, ατμοσφαιρικών ρήπων και ιδιαίτερα του διοξιδίου του άνθρακα. Επίσης ε, έχουν αρχίσει οι, συζήτηση, οι συζητήσεις και γίνεται πρόοδος και είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε την προοδευτική αυτή πορεία με συγκεκριμένα δράσεις, έτσι ώστε να φτάσουμε το ταχύτερο δυνατόν σε μία συμφωνία μεταξύ κρατών μελών. Γι' αυτό θα αρχίσουμε και τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς ε, θεωρούμε ότι θα είμαστε μια ανοιχτή προεδρία και θα θέλαμε από κοινού να μπορέσουμε να επιλύσουμε ορισμένα ζητήματα και θέματα που δεν είναι θέματα μόνο της ε, Προεδρίας, αλλά αποτελούν κοινά προβλήματα και κοινό μέλημα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα Ο κύριος Δεκέρσμακερ, ο Ευρωβουλευτής, ο συγκεκριμένος Ευρωβουλευτής, μίλησε για το θέμα της βιοποικιλότητας. Δεν είναι μόνο η περήφανη η Ρουμανία για τα επιτεύγματα της μέσα στα πλαίσια της εκπεριτροπής προεδρίας. Θα πρέπει να είναι κοινό μας έλλειμμα και ε, κοινή πράξη. Να είμαστε υπερήφανοι όλοι, να προστατεύουμε τα είδη, όλα τα είδη, είτε πρόκειται για πανίδα είτε για χλωρίδα. Γιατί όπως είπατε και εσείς υπάρχουν ε, οι είδη που ήδη την χάνουν προς προστασίας όπως τα μεγάλα σαρκοβόρα, δηλαδή οι αρκούδες και οι λύκοι. Έχουμε λοιπόν κοινέ ανησυχίες και θα γίνει συζήτηση και στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος στο Βουκουρέστι σε σχέση με τα μεγάλα σαρκοβόρα. αλλά θα συνδράμει και ο κανονισμός LIFE. Γιατί φυσικά κινούμαστε μέσα στα πλαίσια του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου και το Life είναι το μόνο πλαίσιο για να προωθήσουμε προωθήσουμε μεγαλόπνοα σχέδια στα πλαίσια του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ότι για το live οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς έτσι ώστε κάθε κρατος μέλος να μπορέσει να συνδράμει και να ευεργετηθεί από το LIFE για μικρά και μεγάλα προγράμματα, βιώσιμα προγράμματα. Πέρα από τον κύριο Λίζε, και ο κύριος Χερμπράντι μίλησε για το θέμα της μακροχρόνιας στρατηγικής για τις κλιματικές αλλαγές. Και όπως είπε και ο κύριος Λίζε, αποτελεί κοινό μας μέλημα και ανησυχία. Θα θέλαμε η διάσκεψη του Συμπίου να είναι ένα πρώτο βήμα έτσι ώστε να ε, ε, εγκριθεί αυτή η σφαιρική στρατηγική. Μιλήσατε για στόχους. Η αναθεώρηση των στόχων μέχρι το 2030 ε, εξαρτάται από τα κράτη-μέλη αποκλειστικά. Και η Ρουμανική Προεδρία θα ασχοληθεί εκ του με το θέμα αυτό έτσι ώστε να μην ξεχαστεί κανένα κράτος μέλος και να προωθήσουμε τις ε, συζητήσεις για να βρούμε τον βέλτιστο δυνατό παρονομαστή. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε σοβαροί για να κινηθούμε προς την κατεύθυνση που επιθυμείτε και εσείς. Η στρατηγική μετά το 2020 για την βιοπικιλότητα θα προωθηθεί άμεσα. Η βιοπικιλότητα ε, είναι ύψη τη σημασίας και για τις επερχόμενες γενιές και έχει μεγάλη σημασία η προστασία της πανίδας και της όριδας ανεξάρτητα από που προερχόμαστε. Η Προεδρία θα προωθήσει την βιοπικιλότητα για την περίοδο μετά το 2020, όπως ανέφερα και στην εισήγησή μου. Θα ήθελα να σας πω ότι οι ανησυχίες μας είναι κοινέ σε σχέση με τα νέα βαρέα όχι κύματα και μιλήσατε για την μακροχρόνια στρατηγική ως προς τις κλιματικές αλλαγές. Θα πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε κοινέ προσπάθειες έτσι ώστε να βρίσκουμε έναν κοινό παρονομαστή. παράλληλα σε σχέση με τις προδιαγραφές ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα για τα νέα βαρέα οχήματα, ε, θα μπορούσα να πω ότι αυτή είναι η ψηφίδα που λείπει από τον κανονισμό οδικών μεταφορών θα πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές σε αντίθεση με την τάση που επικρατεί μέχρι τώρα. Φυσικά έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες αλλά και στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις ελπίζουμε να λάβει τελική μορφή αυτός ο κανονισμός και ελπίζω πριν από το τέλος της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ ε, θα ήθελα να μας έχετε εμπιστοσύνη, μας ενδιαφέρουν άμεσα αυτά τα ζητήματα, θα τα αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα, όπως έγινε και με τις προγενέστερες προεδρίες και θα εντάξουμε και άλλα ζητήματα που θα θέλατε εσείς στο άτυπο, στην άτυπη διάσκεψη ε, για το ε, περιβάλλον στο ΣΥΜΠΗ, ο κύριος Ντένες. Σε σχέση ε, με το ερώτημα του κυρίου Άικχαουτ, σε σχέση με, τα, με το πόσιμο είδωρ, θα ήθελα να σας πω ότι αυτό το θέμα έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα προσπαθήσω να απαντήσω. Η βασική μας προτεραιότητα είναι να φτάσουμε σε ένα εξισορροπημένο συγκεκριμένο κείμενο συμβιβασμού με υψηλό ε, επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας για να ευθυγραμμιστούμε και με τις ποιοτικές προδιαγραφές ως προς το πόσιμο είδωρ να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους και να ενημερώνουμε όπως πρέπει το κοινό. Η διαδικασία διαπραγματεύσεων θα λάβει υπόψη φυσικά και τις γνωμοδοτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ε, Ωραία. Ακολουθεί ο δεύτερος γύρος. Ένα λεπτό έκαστος. Η κυρία Γκροστέτ πρώτη. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο υπουργούς και να επανέλθω λίγο σε μια πληροφορία που μας δώσατε χωρίς λεπτομέρειες, τις ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές. Εδώ τώρα είναι στο σταυροδρόμιο ανάμεσα στο περιβάλλον και την δημόσια υγεία. Το κοινοβούλιο μας έχει εγκρίνει στιβαρά ε, κριτήρια ε, στα βιοκτώνα και στα ε, φυτοφάρμακα για την ταυτοποίηση αυτών των ενδοκρινικών διαταρακτών. Τώρα θα πρέπει να γίνει αυτό εγκάρσια για άλλους τομείς και άλλα είδη προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας κατέθεσε μια στρατηγική που πηγαίνει δεν μένει προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά στερείται συγκεκριμένων άμεσα εφαρμοστών ε, μέτρων. Γιατί υπάρχει έκθεση του πληθυσμού των συμπολιτών μας σε αυτές τις ε, επιβλαβείς ουσίες. Ε, τι σκοπεύει να κάνει η Προεδρία για να προχωρήσει πιο γρήγορα ε, και πιο μακριά. Για το κλίμα επίση ένα τελευταίο. Θέλω να αφαιρθώ στη φορολογία ε, που αφορά την μετάβαση ε, σε μια νέα οικολογική φάση. Είναι λεπτό θέμα, αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να εγγράφεται σε μια γενικότερη στρατηγική για την προστασία του κλίματος και θα σας παρακαλούσα να μας πείτε τις θέσεις σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπράναν. Ε, thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις, ε, λέει ο κύριος Μπράνεν μία για κάθε υπουργό. Προ την Υπουργό Περιβάλλοντο η πρώτη. Και εσεί πολιτικό είστε και εγώ πολιτικό και όλοι εδώ στην Επιτροπή μα πολιτικοί είμαστε. Και επίση γνωρίζουμε ότι είναι και περιορισμένο ο αριθμό των προτεραιοτήτων που μπορεί να έχει μια Προεδρία. Γιατί όταν έχει 73, εκφύσεω δεν είναι προτεραιότητα. Τέσσερι είναι οι προτεραιότητέ σα. Καμία ε, δεν έχει σχέση με την κλιματική αλλαγή ε, Μήπω δεν είναι προτεραιότητά σας, ανησυχώ λίγο και μπορείτε να με καθησυχάσετε ότι όντω είναι. Και επόμενη ερώτηση προς τον Υπουργό Δασών και Υδάτων. Τα, τα δάση ε, συνήθως υποβιβάζονται ε, και μπαίνουν στη γεωργία ή ε, στην ανάπτυξη πέθρου. Αλλά τώρα ε, αποκτούν σημασία ε, σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, γιατί η κάλυψη που έχουμε, η δασοκάλυψη, ε, απορροφάει το 10% του διοξιδίου του άνθρακας. Και τι γίνεται με το ξύλο, όταν το κέμε γίνεται βιομάζα και βλέπουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί η χρήση βιομάζας και μετά χάνεται. Αν όμως το χρησιμοποιήσουμε για τις οικοδομές και αντικαταστήσουμε με το τσιμέντο ε, και φτιάχνουμε ξύλινα σπίτια, ε, θα ε, συνεισφέρουμε στην καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής, γιατί το τσιμέντο και στην παραγωγή του παράγει διοξίδιο του άνθρακα, ενώ όταν είναι ξύλινες οι κατασκευές απορροφούν και διοξίδιο του άνθρακα. Ε, στο μέλλον οι δασοκομεία και τα δάση γενικά θα έχουν πολύ πιο πρωταγωνιστικό ρόλο, κυρίως στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χόισλινγκ. Πολύ συγκεκριμένα έχω μια ερώτηση, διότι η Προεδρία προφανώς πάντα είναι πιο εκτεθειμένη και προβεβλημένη και εκτός της Ένωσης και μπορεί να ξέρετε αυτή την έκθεση από ε, την ε, Euronature που λέει εκτός ελέγχου ότι είναι πολύ ωραία ε, τα δάση και τα, η εθνική δρυμή και τα πάρκα τα οποία καταστρέφονται από την παράνομη καταπάτηση αλλά και από καμία φορά από την εγκεκριμένη από το κράτος. Τι γίνεται με την αξιοπιστία σας. Δεν θα πρέπει να... Ε, ε, μιλάτε για την οδηγία ΕΛΟΚ που θέλετε να την ε, επιβάλλετε παντού. Αλλά βλέπουμε τι γίνεται στη χώρα σας, βλέπουμε τι γίνεται και στη Βρασιλία. Ε, τον κύριο Μπολζονάρο. αλλά όταν πρόκειται για τα δικά μας δάση, τι κάνουμε για να διαφυλάξουμε. Είναι 200.000 εκτάρια προστατευόμενων δασών. Τι κάνετε γι' αυτά. Το Συμβούλιο έχει κάνει τις προτάσεις ε, για την ε, γεωργική πολιτική και δεν, δεν δίνεται μεγάλη προσοχή στη σύνδεση των γεωργικών κονδυλίων με ε, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. Θεωρείτε τέσσερι τις προτάσεις αυτές όπως έχουν κατατεθεί ή μήπως πρέπει να γίνει τίποτα διαφορετικό. Πρόεδρος, χωρίς μικρόφωνο. Okay. Uh... Καλώς. Ο κύριος Ντόρφμαν. Vorsitzende. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ε, που μου δίνετε και χρόνο γόρευσης. Κύριε Υπουργέ, προηγουμένως ε, μιλήσατε μιλήσατε για τα μεγάλα σαρκοβόρα σε σχέση με την ε, βιοπικιλότητα. Λύκους, σαρκούδες και λίγκες. Ε, ε, στη χώρα σας ε, υπάρχουν πολλά σαρκοφάγα ε, μεγάλα. Μπορεί κανείς τώρα να το δει το θέμα αυτό από πλευράς βιοπικιλότητας με διαφορετικό τρόπο. Στο μεταξύ, έχουμε 2.000 αυτό δεν είναι βιοπικιλότητα. Ε, δεν μπορεί να υπάρξει προβατοτροφία σε μεγάλες εκτάσεις γιατί έχουμε πήξει στο λύκο. Ε, ε, τι σχέση έχει πια αυτό με τη βιοπικιλότητα. Έχουν ρημάξει τα πρόβατα. Θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο και τη διαχείριση του λύκου ή αυτών των ειδών για να υπάρξει μια λογική συνύπαρξη μεγάλων σαρκοβόρων από την άλλη και γεωργίας και εκτινοτροφίας από την ε, από τη μια και γεωργίας και εκτινοτροφίας από την άλλη. Και δεν αρκούν τα προστατευτικά μέσα, χρειάζεται και παρέμβαση στον πληθυσμό των ζώων αυτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι τα κράτη έχουν αρκετή ευελιξία και ελευθερία κινήσεων έχετε λάβει και έγγραφα ε, καθοδήγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως που περιορίζει αυτή τη διακριτική ευκαιρία των κρατών. Προτίθεστε να αναλάβετε δράση εκεί ή νομίζετε ότι η κατάσταση που επικρατεί τώρα είναι εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σέρμπου. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σας καλωσορίζω καταρχήν κύριε Υπουργή και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Κυρία Καβριλέσκου, πέρσι ήμουν εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο υπέρ του περιβάλλοντος. Αντιμετωπίσαμε σωρία προβλημάτων και φτάσαμε σε ολέθρια αποτελέσματα σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής. Δεν υπήρχε καμία συνοχή με άλλες πολιτικές. Επίσης δεν υπήρχε σωστή χρηματοδότηση των προγραμμάτων. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο κατά τη διάρκεια της Ρουμανικής Προεδρίας θα, θα ασχοληθείτε με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο υπέρ του περιβάλλοντος και με ποιο τρόπο. Ο κύριος Φλόρεντς. Ναι, κυρία Προεδρεύουσα, κύριε Προεδρεύον. Ε, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούω και είναι και παιδιακά. είστε η εξικοστή και τελευταία προεδρία που ζω. Και αυτά τα 30 τελευταία χρόνια έχω ζήσει πάρα πολλά από παρουσιάσεις και έχω ρωτήσει πάρα πολλούς από τους προκατόχους σας. Πώς θα τα υλοποιήσετε όλα αυτά, γιατί πάντα είστε ε, στην πρώτη γραμμή και δεν χρειάζεται να πάω στη Ρουμανία, μπορώ να μείνω και στη Γερμανία για να τα δω αυτά. Είμαι και Γερμανός. Πολύ ε, αξιέπαινο και ωραίο αυτό που λέτε, ότι θέλετε να ασχοληθείτε με τα ύδατα. Αν δείτε όμως την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, μετά από 25 χρόνια δεν την έχουμε εφαρμόσει. Και σας προειδοποιώ, ε, υπάρχουν διάφορα τεχνάσματα και τα έχει δακτυλουργεί στις διάφορες προεδρίες ε, για να κάνουν διάφορες αλχημίες και να εφεύρουν διάφορους τρόπους να παρακάμψουν την ε, νομοθεσία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία αλλά και προσοχή. Δεν ξέρω, μπορεί κάπου κάποια στιγμή να το παρακάναμε. Δεν το αποκλείω καθόλου στην νομοθεσία, οπότε τα κράτη-μέλη να μην τα εφαρμόζουν γιατί είναι τόσο αυστηρά. Αν δείτε όλες αυτές τις οδηγίες των τελευταίων ετών και πώς αυτές μεταφέρονται και εφαρμόζονται, Ούτε το πρωί δεν θα πηγαίνει κάτω ούτε το πρωινό σας. Παρακαλώ προσοχή και αυστηρότητα να δείξετε. Thank you very much. Uh, Mr. Zani. Κύριο Τζάνι. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για την ε, ευκαιρία που μου δίνετε. Μιλήσατε για αυτά τα μεγάλα ε, αρπακτικά για τα σαρκοβόρα και ούτω καθεξής. Εγώ είμαι Ούγγρος Ευρωβουλευτής, είμαστε μια γειτονική χώρα και θα ήθελα να σας ζητήσω ε, να σας ευχαριστήσω καταρχήν και έχετε προσεγγίσει αυτό το θέμα πολύ καλά. Το κάνατε πολύ προσεκτικά, αν και ε, γνωρίζω ότι η διάσκεψη αυτή θα αποτελέσει μια μεγάλη Καλη πρόκληση. Έχετε συγκεκριμένα προγράμματα. Εάν υπάρχουν ευφυείς τεχνολογίες ε, που να είναι διαθέσιμες, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν υπ' αυτή την έννοια για τη, για τη διαχείριση αυτού του ζητήματος. θέλετε να χρησιμοποιήσετε το λόγο και πάλι. That's very tempting, Chair, but I'll forego that opportunity. Ο κύριος Μπράνεν, ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσω αυτή τη δυνατότητα. Ωραία. Λίγη και ο δεύτερος ε, γύρος ε, ερωτήσεων. Ε, μπορείτε να απαντήσετε ρωτήσετε εσείς πρώτα κυρία Υπουργέ και μετά και ο κύριος Ντένες θα μπορούσε να ε, συμπληρώσει. Κυρία Γκροστέτ, το θέμα των ενδοκρινικών διαταρακτών θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Γιατί αν σκεφτούμε τους χημικούς παράγοντες καταλαβαίνουμε ότι το θέμα αυτό χρήζει διαχείρισης για την ανθρώπινη υγεία και γι' αυτό πρότεινα μία συζήτηση στο, στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος του δικτύου για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Το θέμα αυτό θα πρέπει να το δούμε από κοινού με το Συμβούλιο Υπουργών Υγείας. Θα πρέπει λοιπόν να βασιστούμε σε επιστημονικά δεδομένα, καθώς και στις παρατηρήσεις και διαγνώσεις των καταναλωτών, καθώς και στις ε, τελευταίες ανακοινώσεις της Επιτροπής. Γι' αυτό αποφασίσαμε να γίνει αυτή η συζήτηση και και είμαι πεπισμένη ότι θα φτάσουμε και σε αυτά συμπεράσματα κατά την Προεδρία μας. Αναφερθήκατε επίσης στον έλεγχο, στους ελέγχους σε σχέση με τις κλιματικές Γι' αυτό απάντησα και στον κύριο Λίζ προηγουμένως όταν μιλήσαμε για την στρατηγική των κλιματικών αλλαγών. Θα θέλαμε να μην ε, μιλάμε ε, μόνο στο Συμβουλίο Υπουργών Περιβάλλοντος, αλλά και ε, αγροτικής οικονομίας, ανταγωνιστικότητας, αλλά και οικονομικών. Δηλαδή και μέσα στα πλαίσια του ΕΚΟΦΗΝ να φτάσουμε σε ένα μέτρο σύγκρισης και μέτρο αποτίμησης Κύριε Μπράνεν, όταν μιλήσαμε για τις προτεραιότητες μας και βάλαμε πρώτα τις κλιματικές αλλαγές, δεν το κάναμε τυχαία. Ε, δείτε, μιλήσαμε και για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες που έχουν είναι άμεση συνάφεια με το θέμα των κλιματικών αλλαγών. Θα πρέπει να βασιστούμε στη Συμφωνία του Παρισιού και να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα συμπεράσματα της διάσκεψης. Επειδή μιλήσατε και για τα μεγάλα σαρκοφάγα και το έθιξαν αυτό δύο ευρωβουλευτές, ε, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Τζάνι, και επειδή θα πρέπει να υπάρχει προστασία αυτών των ειδών, θα πρέπει να δούμε έμπρακτα τι μπορούμε να κάνουμε. Άρα δεν είναι καθόλου τυχαίο το θέμα ότι τα μεγάλα σαρκοβόρα τα εντάξαμε στο, συμβούλιο, ε, στο Υπουργικό Συμβούλιο Περιβάλλοντος για να δούμε τι ακριβώς αντιμετωπίζουμε και τι μπορούμε να τροποποιήσουμε καθώς και ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε ε, αυτές οι μετακινήσεις των ε, σαρκοβόρων, καθώς και ο πολλαπλασιασμός τους ε, που μας οδηγεί. Θα θέλαμε ε, να πούμε στον κύριο Μπράνεν ότι θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε. Στη διάσκεψη του Βουκουρεστίου για τα μεγάλα σαρκοβόρα θα φτάσουμε σε αυτά συμπεράσματα, πιστεύω, στο ύψος των προσδοκιών μας. Η κυρία Σέρμπου μας ε, μίλησε για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο υπέρ του περιβάλλοντος. Θα ήθελα να πω ότι μέσα στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος από το 7ο πρόγραμμα δράσης, στο τέλος της θητείας μας και με βάση τις εξελίξεις, όταν θα έχουμε δηλαδή και τα δεδομένα από την Κομισιόν, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα θέλαμε να συνεχίσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις γιατί το θέμα αυτό συνδέεται άμεσα με τις οδηγίες υπέρ του περιβάλλοντος και την εφαρμογή τους. Ασχολούμαστε και με το θέμα της ε, υγείας, αλλά θα έπρεπε να μας απασχολήσει και η αγροτική οικονομία και η ανταγωνιστικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος δεν ε, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Ο κύριος ε, Πρέναν υπέβαλε μία ερώτηση σε σχέση με τη σημασία της ε, δασοκομείας για την απορρόφηση διοξιδίου του άνθρακα και με βάση και τις ε, κλιματικές αλλαγές θα ήθελα να σας ε, τονίσω ότι έχουμε, έχουμε γνώση της σημασίας των δασών στην απορρόφηση του διοξιδίου του άνθρακα. Προσπαθούμε να έχουμε μία σωστή διαχείριση για την ε, μείωση μείωση των εκπομπών που οδηγούν στις κλιματικές αλλαγές. Ο κύριος Χόισλινγκ μίλησε για την κατάσταση στα ε, ΜΜΕ, γιατί φυσικά ε, υπάρχει μία ε, ε, ε, απόκληση της άποψης του κοινού σε σχέση με αυτά που προβλέπει ένα νομοθετικό πλαίσιο και εδώ μιλώ για τις δασοκομικές εκτάσεις που βρίσκονται υπό ιδιωτικό καθεστώς. Υπάρχουν, υπάρχει βέβαια ένα εθνικό σχέδιο που απαγορεύει τις παράνομες ε, υλοτομίες όπου συμμετέχει και η αστυνομία και η, ε, και φυσικά οι συγκεκριμένες αρχές επίβλεψης των δασών για να αντιμετωπίσουν η παράνομη υλοτόμηση. Κύριε Φλόρεν, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Η, οδηγία για τα υδατά για τα είδατα είναι πολύ σημαντική, είναι και πολύ φιλόδοξη, αλλά θα πρέπει να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την πορεία της να υπάρχει σωστή εποπτεία. Δεν θέλουμε να μειώσουμε τους στόχους μας, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντιπρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις απαντήσεις και για την εισήγηση σας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και σίγουρα θα τα ξαναπούμε μέσα στα πλαίσια του τρέχοντος εξαμήνου. Ε, σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Κλείνει αυτό το θέμα να αφήσουμε αφήσουμε τους υπουργούς να αποχωρήσουν και θα συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη. Μια έκτακτη συνεδρίαση μας θα λάβει χώρα στο Στρασβούργο στις 14 Φεβρουαρίου 8.30 έως 10.30 πρώμη συμβρία για να ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση για τις προτάσεις στρατηγικών σχεδίων για την κοινή αγροτική πολιτική. Το προσχέδιο μερίσιας διάταξης θα κυκλοφορήσει εν ευθέτω χρόνο. Δεύτερον, κατόπιν τη υιοθέτηση τη Επιτροπή της Έκθεση Επιτροπή ε, Πέση, Επιτροπή Αδειοδότηση Παρασιτοκτόνων, η Κριστίνα Μάλμρο και η Νόρα Χάν Κάμπερ επανέρχονται στη γραμματεία τη ΕΜΒΗ. Καλώ ήρθατε. Έχουμε 20, 20 γλώσσες διερμηνία σήμερα και όπω ε, ε, η συνεδρίαση μεταδίδεται μέσω ε, ίντερνετ ζωντανά και θα είναι διαθέσιμη και στο e-meeting. Έχετε επίσης πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων στο φάκελό σας των έξι προηγούμενων συνεδριάσεων Αν δεν έχετε αντιρρήσει μέχρι το τέλος της θα θεωρήσω ότι εγκρίνονται. Τώρα, για τις ε, διοργανικές διαπραγματεύσεις που διεξάγονται αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την αναδιατύπωση ε, της, ε, του κανονισμού για τους επίμονους οργανικούς, τους ε, έμμονους οργανικούς ρήπους. 18 ε, Δεκεμβρίου έγινε, ε, λόγο, έγινε ο δεύτερος τριμερής διάλογος. δεν καταλήξαμε σε συμφωνία. δεν καταλήξαμε συμβιβασμό για το, το βασικό πολιτικό θέμα που αφορά τα όρια συγκέντρωση των ουσιών των παρατημάτων 4 και 5 και τον τρόπο με τον οποίο αυτά θα τροποποιούνται. Κόμμα πρόταση κομισιών που δεν τροποποιήθηκε από το Κοινοβούλιο προβλέπει αυτά τα όρια να καθορίζονται στα παρατήματα 4 και 5 και σε κατεξοδότηση πράξης για την αλλαγή του Όμω, τους. Όμως το Συμβούλιο επιθυμεί να χρησιμοποιούνται πράξεις, εφαρμοστικές πράξεις. Ε, θα γίνει άλλος ένας τριμμένος διάλογος τον Ιανουάριο, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε. Σε ό,τι αφορά ε, τις προδιαγραφές για τα διοξίδια του άνθρακα στα βαρέα οχήματα, πρώτος τριμμένος διάλογος ε, έλαβε στις 8 Ιανουαρίου, πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ο στόχος ήταν ε, οι συνεισηγητές ε, να ε, στείλουν όσο το περισσότερα θέματα στους τεχνικούς εμπειρογνώμονες και να εξετάσουν τις τροπολογίες προκειμένου να δοθούν περισσότερες διευκρινήσεις εν ώψη του επόμενου διαλόγου που θα γίνει αύριο 22 Ιανουαρίου. Πρόγραμμα για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή LIFE Ο πρώτος τριμερής διάλογος για το LIFE έλαβε χώρα σε 9 Ιανουαρίου Ε, παρουσιάσαμε τις θέσεις μας, έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τα βασικά θέματα. Οι συζητήσεις κατέριξαν ότι και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν παρόμοια προσέγγιση για ένα, αριθμό, για θεμάτων εκτός ιδιαίτερως για τους στόχους των προγράμματος, θέματα χρηματοδότησης, ε, συντελεστές χρηματοδότησης, γεωγραφική ισορροπία και τις διατάξεις ειδικέ με την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας μέσω ε, πράξης, ε, ε πράξης ή πράξεων εφαρμοστή. Θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση στο επόμενο, στην επόμενη συνεδρίαση 7 Φεβρουαρίου. Διαφάνεια και βιωσιμότητα ε, στην ε, εξορρόηση κινδύνου στην ε, τροφιμική αλυσίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτος τριμμένης διάλογος Δευτέρα 14 Ιανουαρίου. Ε, παρουσιάστηκαν οι θέσεις σε κατέρωθεν Ορισμένα θέματα παραπέμφθηκαν στους εμπειρογνώμονες. Ε, ο χρόνος πιέζει προκειμένου να κλείσει το θέμα, οπότε συμφωνήσαμε τα πολιτικά θέματα να συζητηθούν και σε τεχνικό επίπεδο προκειμένου να προετοιμαστεί η πολιτική συζήτηση. Δεύτερη συνεδρία πολιτικού διαλόγου την 5η 24 Ιανουαρίου. Αυτά σε σχέση με τον διοργανικό διάλογο. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Ε, τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας. ο κ. Πιέκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Τα τελευταία χρόνια πρέπει να σας πω ε, είναι πολύ μεγάλο θέμα και απασχολεί την κοινή γνώμη αυτή η αλλαγή της ώρας ε, και διάφορα επαγγέλματα γιατροί, αγρότες, ε, εργαζόμενοι στις μεταφορές προβληματίζονται. Κανονικά η κανονική ώρα στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η χειμερινή ώρα. Αυτή είναι για η βασική ώρα. Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση ε, ε, δέχτηκα την πρώτη πρόταση αυτή, την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι αποτέλεσμα ε, της γνώμης πολλών Ευρωπαίων, χιλιάδων Ευρωπαίων και αρκετών Ευρωβουλευτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε μία απόφαση να αναθεωρηθεί η αλλαγή της ώρας. Της θερινής όμως. Να αλλάζει από χειμερινή σε θερινή. Θα γίνει μια αξιολόγηση αν χρειάζεται να τερματιστεί αυτή η αλλαγή, όχι. Και η δική μας Επιτροπή, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, σε ένα έγγραφο που ασχολείται και με θέματα περιβάλλοντος αλλά και με τη δημόσια υγεία, πώς επηρεάζει η αλλαγή της ώρας τους πολίτες και γενικά τη ζωή στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να πούμε ότι ε, ασκούνται πιέσεις από διάφορες πλευρές και οι ιατροί αντιδρούν, υπάρχουν θέματα υγείας πολύ σημαντικά. Είναι ένα ολόκληρο φάσμα λοιπόν αυτό που, των προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την αλλαγή της ώρας. Μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα περισσότερο έχουμε επιπτώσεις λίγες μέρες με την αλλαγή της ώρας, αλλά ορισμένες φορές είναι και μακροπρόθεσμες. Η ε, αλλαγή της ώρας λοιπόν έχει και θετικές πτυχές και αρνητικές. Επηρέαζει αρνητικά του τους βιορυθμούς το βιολογικό ρολόι μας. Αλλά και αυτό ακόμα είναι αντικείμενο μελέτης, δεν έχουν καταλήξει οι ειδικοί για το πώς προσαρμόζεται ο ανθρώπινος οργανισμός στην αλλαγή της ώρας. Επίσης προσπάθησα να λάβω υπόψη μου τις διάφορες πηγές, επιστημονική βιβλιογραφία κτλ. που κάνουν λόγο ε, για την ευημερία του πληθυσμού στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν υπόψη και τα επιστημονικά δεδομένα. Έχει γίνει βρία διαβούλευση για το θέμα αυτό, όχι μόνο δημόσια, για την αλλαγή της ώρας, για να εγκαταλείπουμε τη χειμερινή και να περνάμε στη θερινή ώρα. Ε, ε, δεν ήταν μόνο διαβούλευση λοιπόν αυτή που έγινε, γίνανε πολλές μελέτες, στατιστικές κτλ. Πώς επηρεάζει τους πολίτες. Ας πούμε υπάρχει Υπάρχει μια στατιστική που λέει ότι αυξάνονται τα εμφράγματα του μυοκαρδίου ε, και αυτό έχει σχέση με την αλλαγή της ώρας ή αυξάνονται οι αυτοκτονίες. Ο κόσμος είναι πιο δυστυχισμένος από τη ζωή του. Ή γίνονται διάφορα δυστυχήματα στην κυκλοφορία στους δρόμους ε, όταν αλλάζει η ώρα, ανοιχτό αν είναι νωρίτερα κτλ. Ε, αυτό επηρεάζει ψυχολογικά τον κόσμο. Επίσης βασίστηκα και σε αναλύσεις που έγιναν ε, ως προς το πώς επηρεάζει η αλλαγή της ώρας στον ανθρώπινο οργανισμό. Όπως σας είπα λοιπόν, είναι ευρύτατο το φάσμα αυτό των προβλημάτων. Ξέρω ότι είναι της μόδας ε, να κατηγορούμε την αλλαγή της ώρας και να θεωρούμε αρνητική μεταξύ άλλων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της κυρίως κάνει λόγο για τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και καλό θα ήταν να το κοιτάξουμε αυτό το θέμα. Ε, και να αφήσουμε ε, όμως τη διακριτική ευχέρεια στα κράτη-μέλη. Ξέρετε ότι αν αρχίσουμε από την Εστονία, τη Λιθουανία, τη Λετωνία και φτάσουμε στην Πορτογαλία, δεν έχουμε παντού την ίδια ώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολλές ε, διαφορές μέχρι δύο ώρες. Συμφωνώ με την ανάλυση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιτροπής ότι υπάρχουν επιπτώσεις για τη δημοσία υγεία. Αλλά ας αφήσουμε τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν. Να πάρει το κάθε κράτος τη δική του απόφαση αν θα εναρμονιστούν οι αποφάσεις τώρα με βάση όλα τα επιχειρήματα και όλες τις φωνές που ακούγονται. Δεν είναι καθόλου εύκολο το θέμα αυτό. έτσι, ε, ε δίστανται οι απόψεις η Πορτογαλία, η Εστονία, η Λετωνία, η Γερμανία μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη. Εμείς θα πρέπει να δείξουμε καλή θέληση και να τα συζητάμε όλα αυτά τα θέματα. Αλλά είναι ένα ζήτημα που απασχολεί δεκαετίες ολόκληρες στον κόσμο και προσπαθούμε να το λύσουμε. πολλοί κόσμος έχει συνηθίσει να αλλάζει η ώρα, αλλά οι νέοι αντιδρούν. Ε, υπάρχουν και άλλα ζητήματα, οι μεταφορές, οι αερομεταφορές, η γεωργία, αλλά δεν είναι πάντα επαρκή τα στοιχεία τα εμπειρικά για να μπορέσουμε ε, να καταλήξουμε κάπου μόνο σήμαντα και κατηγορηματικά. Ας αφήσουμε στα χέρια των κρατών μελών. Αυτά προ... από μένα. Ευχαριστώ. Ποιος άλλος θα ήθελε το λόγο? Ο κ. Λίζα λείπει, έρχεται αυτή τη στιγμή, έχω μάθει. Και ο κύριος Ντάντς επίσης. Να δώσω το λόγο στην Κομισιόν εδώ μεταξύ. Να κάνει τα σχόλιά της και μετά... Α, ε, αν οι άλλοι δύο σκιοσηγητές στήξουν κάποιο θέμα που σας ενδιαφέρει, σας ξαναδίνω το λόγο. Καλώς απόγευμα. Ονομάζομαι Πίτερ De ε, Έχω συναντήσει με τον εισηγητή και μπορώ να είμαι πολύ σύντομος γιατί χαιρόμαστε για την ε, έκθεση της Επιτροπής. Έχουμε λάβει υπόψη τη γνώμη του κ. Πίσα. Προτείνει την ε, αναβολή εφαρμογή μέχρι το 2020, δεδομένη τη κατάσταση του Συμβούλιο, φαίνεται λογική αυτή η πρόταση. Η γνωμοδότησή του είναι στην, στο ίδιο μικρό με τις δικές μας προτάσεις, οπότε του ευχόμαστε καλή τύχη. Περιμένουμε την τελική συνολική γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου και εντωμεταξύ θα είμαστε στη διάθεσή σας. Okay, thank you very much. Πρόεδρος. Ωραία. Κύριε Πιέκα. Ευχαριστώ. Ε, θα θέλαμε προφανώς η, η αλλαγή να γίνει το συντομότερο δυνατό, αλλά δεν νομίζουμε ότι αυτό είναι δυνατό, διότι υπάρχουν κάποιες διαδικασίες στις οποίες πρέπει να σεβαστούμε, υπάρχουν διάφορες επιτροπές οι οποίες έχουν γνωμοδοτήσει για το ζήτημα και μετά έχουμε και τρία όργανα, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Κομισιόν. Οπότε λογικό είναι να αφήσουμε το θέμα αυτό, να αφήσουμε την εφαρμογή για το 2021. Να ομολογώ όμως ότι εγώ προσωπικά θα προτιμούσα να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα. Δυστυχώς όμως αυτό δεν γίνεται. Okay, then, thank you very much. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Ε, ολοκληρώνεται λοιπόν και το θέμα αυτό. Προθεσμία για την κατάθεση απολογιών 25 Ιανουαρίου και ελπίζουμε να ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας το Φλεβάρι 20 και 21 του μηνός. Και προχωρούμε τώρα στους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Έχουμε τέσσερις αντιρρήσεις σε κοινή συζήτηση. Καλώ τους συνεισηγητές να λάβουν το λόγο. Είναι εδώ ο κύριος Μπάρτ Στάς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι αγαπητοί παρόντες εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μαζί με μέλη από όλες τις άλλες πολιτικές ομάδες ε, καταθέσαμε μία αντίρρηση για την κυκλοφορία στην αγορά ε, τεσσάρων νέων ε, κοιλιών, ε, ελαιοκράμβη, αραβόσιτο, ε, δύο είδη αραβοσίτου και βαμβάκι. Ε, δεν θα σας παρουσιάσω όλες τις αντιρρήσεις. Έχουμε ψηφίσμα, ψηφίσματα τα οποία θα εγκρίνουμε προσεχώς σε λίγο, αν πάνε και στην Ολομέλεια, θα καταφέρουμε ε, ε, να έχουμε περάσει 31 αντιρρήσεις ε, κατά τη διάρκεια της παρούσης θητείας και οι πλειοψηφίες στην Ολομέλεια είναι γύρω στα 2 τρίτα, κινούνται πάντα γύρω στο 66%. Και αυτό πραγματικά είναι πολύ ε, απορίας άξιο, γιατί ερχόμαστε και διαπιστώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να εγκρίνει ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς για τρόφιμα και ζωοτροφές, παρόλο που ξέρουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν τρελαίνονται κιόλας για αυτά και στο Συμβούλιο Υπουργών δεν υπάρχει ειδική ενισχυμένη πλειοψηφία για να κυκλοφορήσουν στην αγορά αυτές οι γενετικά τροποποιημένες ποικιλίε ε, τροφίμων και ζωοτροφών. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί κατεβάζει συνέχεια τέτοιες προτάσεις. Και μάλιστα όταν ο τύπος ε, κοιτάει αλλού, ξέρω εγώ, θερινές διακοπές ή χριστουγεννιάτικες διακοπές, ε, πολύ στοχευμένα και πολύ περίεργα μου φαίνονται όλα αυτά. Δεν θα μιλήσω για το δημοκρατικό έλλειμμα, αλλά να κάνω κάποιες ερωτήσεις επί της ουσίας ε, στον πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτον, διάφορα μεταλλαγμένα φυτά ε, εδώ ε, ε, είναι αντεκτικά στη γλυφοσάτη που, που είναι τοξική και που απαγορεύεται η χρήση. Κυρίως το ελαιοκράμβι και το βαμβάκι αφορά αυτό και τη γλυφοσυνάτη ε, και μάλιστα αυξάνεται η αντίσταση τους και αυξάνεται και η δόση ε, της ουσίας αυτής σε σχέση με ε, τις συμβατικές ε, καλλιέργειες ε, και βάμβακος. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για κατάλοιπα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει πει σε προηγούμενες συζητήσεις ε, ότι ε, δεν υπάρχει πρόβλημα για τους πολίτες γιατί ε, ε, μετράμε ε, τα μέγιστα κατάλοιπα που επιτρέπονται. Για το επόμενο διάστημα, 2019 2021, όμως δεν είναι υποχρεωμένα τα κράτη-μέλη να μετρούν τα κατάλοιπα της γλυφοσυνάτης. Ρωτώ λοιπόν, ε, πώς μπορεί να μας εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη βεβαιότητά της. Ότι οι πολίτες ή τα παραγωγικά ζωά δεν θα είναι εκτεθειμένα ε, στις υψηλές δόσεις γλυφοσυνάτης. Γιατί δεν είναι και υποχρεωτική πλέον η έλεγχη από τα κράτη-μέλη. Η αρχή της προφύλαξης δεν θα επέβαλε ε, να απαγορευτεί η εισαγωγή όλων αυτών των ε, γενετικά τροποποιημένων φυτών που εμφανίζουν υψηλή αντίσταση σε όλα αυτά τα τοξικά φυτοφάρμακα τα οποία έτσι κι αλλιώς απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, αξιόπιστες επιστημονικές ε, πληροφορίες λένε ότι το βαμβάκι ε, έχει μεγάλες ε, συγκεντρώσεις της τοξίνης οξυπόλ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ε, Γκοσιμπόλ, συγγνώμη, για το βαμβάκι που είτε ως πλακούντας στις ζωοτροφές και το βαμβακέλαιο. Τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με αυτά. Μια μελέτη του 2004 αναφέρει σε σχέση με την ύπαρξη ότι υπάρχουν προβλήματα ε, αναπαραγωγής ανδρών και γυναικών ε, και μεγάλες οικονομικές απώλειες στους κτηνοτρόφους αλλά και ότι επηρεάζεται αρνητικά το ανοσοποιητικό και είναι πιο ευάλωτος ο πληθυσμός σε λοιμώξεις. Ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς ε, διαχειριζόμαστε τον κίνδυνο και γιατί δεν το έχετε αναθέσει στην ΕΦΣΑ. Ε, το έργο της ΕΦΣΑ σας αρκεί σε αυτή την ε, υπόθεση. Και τελευταίο το γενετικά τροποποιημένο βαμβάκι που μας απασχολεί. Εκτός αυτού, αντίσταται και στα ε, αντιβιωτικά. Ε, έχει ε, δι, στρεπτομικίνη, νεομικίνη και κάναμικίνη. Έχει κάποιους δείκτες που στα προϊόντα αυτά ε, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έχουν ταξινοποιηθεί ε, ως υψηλής ε, σπουδαιότητας. Εδώ όμως το αντίστοιχο πάνελ της ΕΦΣΑ το 2004 έχει μελετήσει αυτά τα γονίδια δείκτες για την αντοχή αντιβιωτικά. Και πού καταλήγει ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αντοχή των ανθρώπων και των ζώων αντίσταση σε κάποια είδη αντιβιωτικών. Ερωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζουμε όλοι ε, ε, ποια είναι η πρόκληση ε, αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος της αντοχής στα αντιβιωτικά. Για ποιο λόγο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εγκριθεί αυτό το γενετικά τροποποιημένο βαμβάκι. Ευχαριστώ. Αυτά τα ολίγα. Thank you very much. Now, on behalf of me. Η κυρία του κυρίου Μπάλας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν έλαβα εγώ εξ του Γκυγιόμ Μπάλας να σας παρουσιάσω την ομοδότηση σοσιαλιστών και δημοκρατών και δεν μπορώ παρά να επαναλάβω. Ε, επανειλημμένα μας έχει ε, απασχολεί σε αυτό το θέμα και δεν είναι 31 ουσίες που ανέφερε. Ε, ο Μπάρτ μίλησε για 31, είναι 32. Έχω μετρήσει μία παραπάνω. Ε, το πρόβλημα ποιο είναι τώρα εδώ με τις αντιρρήσεις αυτές κατά των γενετικά τροποποιημένων ε, οργανισμών. Είναι πολύ απλό να το περιγράψουμε. Όπως και πολλά επιστημονικά τα ανέφερε ο Μπάρτ Στάς, αυτό που μας ε, ανησυχεί μας και μας βασανίζει είναι ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στο Συμβούλιο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει. Η Επιτροπή Προσφυγών το Γενάρη δεν αντέδρασε, δεν πήρε καμία απόφαση για καμία από τις ουσίες αυτές. Το αποτέλεσμα ήταν no opinion. Η χώρα μου, η Γερμανία και στις τέσσερις ψηφοφορίες απήχε. Ε, αυτό είναι πάγια πρακτική εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε δεν μπορούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργούμε σοβαρά και να συνεργαζόμαστε με νόημα. Γι' αυτό χρειάζεται να αναθεωρηθεί αυτή η διαδικασία και κατά τη διάρκεια ακόμα του της δότης θητείας θα ψηφίσει το Κοινοβούλιο της Αλλαγέ. Οι συνάδελφοι της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων έχουν επιληφθεί. Ε, πριν τεθεί σε ισχύει η νέα λοιπόν διαδικασία, κανονικά εμείς δεν θα πρέπει να εγκρίνουμε καμία κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από πλευράς περιβάλλοντος θέλω να τονίσω ένα ακόμα στοιχείο. Σε όλες αυτές τις διαδικασίες έγκρισης πρόκειται για θέματα δημόσιας υγείας. Το ξέρω ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις και διαφορετικές. Ε, αλλά ποτέ δεν μετράμε τις επιπτώσεις ε, στο περιβάλλον, μόνο τη δημόσια υγεία ελέγχουμε. Άρα θα πρέπει να αναθεωρηθούν τα κριτήρια. Το ελπίζουμε και η ομάδα σοσιαλιστών και δημοκρατών ε, συνιστά να εγκρίνουμε τις αντιρρήσεις αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Φλόρεντς. Ευχαριστώ. Και εγώ διαμεσολαβητής είμαι. Να σας πω τι λέει το ΕΛΚ. Στις πρι... τις πρώτες αντιρρήσεις θα υπερψηφίσουμε. Στην τέταρτη που αφορά το γενετικό τροποποιημένο βαμβάκι και τις αντιστάσεις και αντοχή ε, στα αντιβιωτικά κτλ. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε εδώ ότι υπάρχει ανάπτυξη, αντίσταση στα αντιβιωτικά φυσικά ανεπιθύμητη, ε, ειδικά στο στα γονίδια ADD. Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας διαβεβαιώσει ότι ε, αν κυκλοφορήσει στην αγορά αυτό το βαμβάκι δεν θα έχουμε πρόβλημα αύξησης ε, της αντίστασης αντιβιωτικά. Μπορεί να μας εγγυηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί επειδή ασχολούμαι με τη Γεωργία και εγώ ανησυχώ για αυτά τα πράγματα, όπως και άλλοι. Άλλος κανείς. Για να δούμε τι έχει να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Dear members of Parliament. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε πολύ προσεκτικά όλα τα σχόλια. Και θα θέλαμε μία ακόμα φορά να υπογραμμίσουμε ότι είναι υποχρέωσή μας, νομική υποχρέωσή μας, να ακολουθήσουμε τις διαδικασίες που προβλέπονται από την νομοθεσία περί γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. Αυτό μπορώ να σας εγγυηθώ είναι ότι αυτές οι διαδικασίες θα ακολουθηθούν με τη μέγιστη προσοχή. Η ΕΦΣΑ έκανε την αξιολόγηση κινδύνου για όλα αυτά τα προϊόντα και επιβεβαίωσε ε, ότι δεν τίθεται θέμα ασφάλειας. Ακόμα και σε ό,τι αφορά τον, το γονίδιο ε, ε, αντίσταση στα αντιβιωτικά. Η ΕΦΣΑ μας ε, διαβεβαιώνει ότι και, αυτός, και αυτή η πτυχή εξετάστηκε και δεν δημιουργείται πρόβλημα σε σχέση με το συγκεκριμένο οργανισμό. Και ο Στάση έθιξε το θέμα των ε, υπολοιμάτων. Καταρχήν να υπογραμμίσουμε ότι όλα τα φυτά τα οποία εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τηρούν τα όρια της νομοθεσίας περί ε, μέγιστης συγκέντρωσης. Λοιπόν. Και θα πρέπει να ε, αυτό να λαμβάνει υπόψη στα ετήσια σχέδια ελέγχων. Αν τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι αυτού του είδους τα όρια δεν είναι κάτι το επικίνδυνο, μπορούν να μην, να μην τα περιλαμβάνουν στα αιτήσια σχέδιά τους, αλλά η νομοθεσία θα πρέπει να τηρείται. Καταλαβαίνω βέβαια ότι μας ρωτάτε γιατί εξακολουθούμε να εγκρίνουμε ε, γενετικά τροπημένους οργανισμούς. Εγώ θα σας πω ότι ακολουθούμε την νομοθεσία. Ένα κρατός μέλος δεν ψηφίζει ότι παίρνετε κατά, αλλά οι ζωοτροφές εισάγονται για όλες τις χώρες. Οπότε η ερώτηση είναι γιατί δεν παίρνετε θέση. Ε, οι ζωοτροφές αυτές εξακολουθούν να εισάγονται γιατί είναι ασφαλείς και χρησιμοποιούνται. Οπότε υπάρχει ένα θέμα εξάρτησης, αλλά δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας. Το άλλο θέμα έχει σχέση με την απουσία γνωμοδότησης. Όπως γνωρίζετε η Κομισιόν έχει προτείνει την αύξηση, τη βελτίωση της διαφάνειας ε, με συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες την χάνουν διαπραγμάτευση ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή. Μακάρι να συνεχιστούν οι συζητήσεις και να ολοκληρωθούν. Οι αντιρρήσεις για, τις, ε, για τους οργανισμού οργανισμούς δεν μπορούν, μπορούν να είναι πολιτικές, αλλά δεν μπορεί να είναι βασισμένες σε ανησυχίες ότι αφορά την ε, ασφάλεια, διότι η ΕΦΣΑ έχει κάνει την αξιολόγηση κινδύνου. Ακόμα και οι διαδικασίες της ΕΦΣΑ ε, την είχαν διαπραγματεύσει αυτή τη στιγμή, τις παρακολουθούμε. Ε, το μόνο που μπορώ να πω εγώ αυτή τη στιγμή είναι ότι ε, το δικαίωμα ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι περιορισμένο στο κατά πόσον έχουμε υπερβεί τις εκτελεστικές μας εξουσίες, κάτι που δεν έχουμε κάνει. Εμείς αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε την υφιστάμενη νομοθεσία περί γενετικών τροποποιημένων οργανισμών. Προφανώς πάντοτε είμαστε στη διάθεσή σας για επεξηγήσεις, αλλά τα επιχειρήματα τα οποία προβάλλατε σήμερα δεν σχετίζονται ε, και υπερβαίνουν το δικαίωμα ε, ελέγχου ε, κοινοβουλευτικού ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς βασιζόμαστε στην νομοδοτήσεις της ΕΦΣΑ, οι οποία στις συγκεκριμένες περιπτώσεις και στις τέσσερις περιπτώσεις έχει επιβεβαιώσει πως δεν τίθεται θέμα ασφάλειας. Ευχαριστώ. Και νομίζω ότι μπορώ να σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ψηφίσουμε αύριο, συνάδελφοι, ε, για τις αντιρρήσεις αυτές και ε, στη δεύτερη ολομέλεια του Ιανουαρίου. Ε, ψηφοφορίες τώρα έχουμε, αλλά για τις 5 και 20. Οπότε και θα διακόψουμε μέχρι τις 5 και 20. Πείτε κανένα καφέ, κανένα τσαγάκι.